Colleagues, please be seated. Those who would like to leave the chamber, please proceed and do it. Παρακαλώ πολύ καθίστε να προχωρήσουμε. Έχουμε δουλέψει πολύ καλά μέχρι τώρα. Ε, θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως και θα καλωσορίσω ε, τον, ε, τον κύριο Άντρης Πέλτς, τον πρέσβη της, Λετο, της, Λιθουανία, της Λετωνίας, συγγνώμη, ο οποίος ε, έχει από το πρωί παρακολουθήσει, αν δεν κάνω, καλά, αν δεν κάνω λάθος, ε, όλες τις ε, σχετικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου ε, οι οποίες είναι αφιερωμένες ακριβώς στο θέμα της κοινή ε, πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης είναι ε, η αλλαγή του περιβάλλοντος όσον αφορά την άμυνα και την ασφάλεια και το μέλλον της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας πρέπει να σας πω ότι τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ. Είναι ένα περιβάλλον το οποίο τάχιστα τροποποιείται, ε, γιατί η κατάσταση είναι δυναμική, ε, πάρα πολύ δυναμική μάλιστα, και επομένως ε, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και από τη δική μας πλευρά. Έχουμε λοιπόν ε, ε, μαζί μας ε, τον εκπρόσωπο της χώρας, της Λετωνίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε λοιπόν τον λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την δυνατότητα ε, να δούμε τις εξελίξεις καθώς επίσης ε, και τα, τον σχεδιασμό ο οποίος ε, υπάρχει έτσι, σχετικά με την υλοποίηση της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, μέλη, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ξεκινήσω με μία μικρή ε, δήλωση σχετικά με το τι συνέβη τους τελευταίους έξι μήνες, στη διάρκεια δηλαδή της ε, Προεδρίας μας ε, όσον αφορά τα θέματα άμυνας και ασφάλειας στα πλαίσια των ομάδων εργασίας των οποίων είχε την τιμή να προεδρεύει η Λετωνία και βεβαίως μετά μπορείτε να θέσετε και οποιασδήποτε ερωτήσεις. η Λετωνία ξεκίνησε την προεδρία της ε, σε μια κατάσταση ασφάλειας ε, ιδιαίτερα περίπλοκη, ίσως την πιο περίπλοκη μετά από το τέλος του ψυχρού πολέμου, ε, ε, μετά από τα τεκτενόμενα στην Κρυμαία, την προσάρτηση από την Ρωσία και τα λοιπά, έπρεπε να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες προκλήσεις. Επιπλέον, η διονγκούμενη αστάθεια και στην ε, Μέση Ανατολή αλλά και σε πολλές περιοχές ε, της ε, Αφρικής είχε σαν αποτέλεσμα μεγάλα ρεύματα μεταναστών και συγγνώμη ετούντων άσυλων να και προσφύγων να φύγουν από τη Λιβύη, από τη Βόρεια Αφρική αλλά και τη Μέση Ανατολή, Συρία κλπ. προς την Ευρώπη. η Επιτροπή Ασφάλειας αλλά και άλλες ε, ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στον Γενικότερο Μηχανισμό Άμυνας και Ασφάλειας έχουν ε, ασχοληθεί με, το, με τα θέματα αυτά. Το χρονοδιάγραμμα της ε, άμυνας και ασφάλειας και το θεματολόγιο είναι ιδιαίτερα ποικίλο και με μεγάλες μεταπτώσεις. Να σας πω ότι ε, προσπαθήσαμε να, προσπαθούμε κάθε χρόνο να βρούμε τα κυριότερα 10 ε, σημεία ε, για την επόμενη χρονιά και φέτος τα περισσότερα είναι καινούργια ζητήματα. Για όλους αυτούς τους λόγους το θεματολόγιο της άμυνας και της ασφάλειας ε, ασχολείται με πολλά θέματα, αλλά πολύ περισσότερο με την τρομοκρατία και την μετανάστευση. Ε, γι' αυτό ακριβώς ε, αποφάσισαν οι Υπουργοί Άμυνας να δημιουργήσουν μια ναυτική δύναμη αποτροπής για τα μεταναστευτικά κύματα της Μεσογείου κυρίως αργότερα θα συζητήσουμε και για το θέμα αυτό. Εξακολουθούν βεβαίως να παραμένουν με υψηλή προτεραιότητα και για την Λετωνία κυρίως ε, η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, ε, η ε, συνεργασία με τις ε, Ηνωμένε Πολιτείες, ε, η στρατιωτική ικανότητα και ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα αντιμετωπίζεται. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι η επιτυχία όλων αυτών των διεργασιών εξαρτάται από το κατά πόσο ο κυβερνοχώρος είναι και θα εξακολουθήσει να είναι ασφαλής. Επομένως, θελήσαμε να δημιουργήσουμε το πλαίσιο ασφαλούς ε, κυβερνοχώρου ως ε, κύριο συστατικό της ε, κοινή πολιτικής άμυνας ασφάλειας. Στη διάρκεια της Προεδρίας μας διεπροετοιμάσαμε μια, μια διάσκεψη για την προστασία του κυβερνοχώρου όπου συζητήσαμε ακριβώς αυτό το πλαίσιο της κυβερνοασφάλειας. Επίσης, Είχαμε συζητήσεις ε, σχετικά ε, με τη διασύνδεση ανάμεσα στην εξωτερική και την εσωτερική ασφάλεια. Ε, τα ζητήματα αυτά ε, μπήκαν στην ημερήσια διάταξη διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα συζητηθούν και στην στο επερχόμενο Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Σε ορισμένα θέματα έχουν γίνει πρόοδοι, πολλές φορές η πρόοδος είναι μεγαλύτερη σε ορισμένα ζητήματα, σε άλλα λιγότερη. Εν πάση περιπτώσει Έγινε πολλή δουλειά στη διάρκεια της εξάμηνης προεδρίας της ε, Λετωνίας και οδηγηθήκαμε σε καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να προωθήσει ε, τις προσπάθειές της ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει ε, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό. Ε, μεγάλο τμήμα δε αυτού του Συμβουλίου θα αφιερωθεί σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Περισσότερη προσπάθεια και δουλειά θα πρέπει να γίνει για την ανανεωμένη εσωτερική, ε, ε, ε, συγγνώμη, στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα στο οποίο αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία και αναμένουμε ότι η ύπατη εκπρόσωπος θα κάνει μια σχετική παρουσίαση. Αυτό που είναι εξαιρετικά υψηλή σημασία είναι να δούμε την διασύνδεση ανάμεσα στη στρατηγική εσωτερικής και τη στρατηγική εξωτερικής ασφάλειας διότι η, η, τα όρια αυτών των δύο περιοχών γίνονται όλο και πιο ασαφή. Το Δεκέμβριο του 2013 είχαμε καταλήξει στο Συμβούλιο σε διάφορα ε, συμπεράσματα όσον αφορά την ε, ε, ορατότητα, την σαφήνεια και την ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων και αυτά μας οδήγησαν μέχρι τώρα και μέχρι το 2015. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την ΕΝΤΑ, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία υπηρεσία ε, άμυνας ε, και έχει κάνει επομένως συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση απειλών ε, και θα συζητήσετε το πλαίσιο αυτό φέτος. Θεωρούμε ότι η παρούσα ε, κατάσταση της Ευρώπης μας οδηγεί στις προκλήσεις τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και στα διακυβεύματα τα οποία ε, έχουμε. Ε, βεβαίως ε, εμείς στηρίζουμε την μη επικάλυψη προσπαθειών. Τη, λέμε ότι και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν σαφώς περιγραμμένους ρόλους, αλλά θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίζουν κάποια ζητήματα πολύ σημαντικά, όπως ας πούμε αυτό του υβριδικού πολέμου. Όλα τα κράτη τα οποία συμμετέχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στο ε, ΝΑΤΟ έχουν ιδιαίτερο ρόλο να παίξουν. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως θα πρέπει να λαμβάνονται οι ε, πάντα στα πλαίσια της συμπληρωματικότητας και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι δραστηριότητες. Επίσης και κάποιες άλλες πρακτικές δραστηριότητες ανέλαβε η Προεδρία. Ε, ας πούμε ασχολήθηκε με την χρηματοδότηση των ε, ε, κοινών προγραμμάτων όσον αφορά την καταπολέμηση απειλών όπως ας πούμε το Αθήνα, όπως ας πούμε η Αταλάντα, όπως επίσης η αποστολή στο κέρας της Αφρικής ή στο Μαλί. Το σύνολο της χρηματοδότησης είναι περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ ε, τα ε, ε, οποία αφορούν και τις, τους στρατιώτες και την υποστήριξή τους. Θα ήθελα να υπογραμμίσω σύντομα τους τομείς τους οποίους έχουμε διαπιστώσει κάποια πρόοδο. Πρώτον, στη διάρκεια της Λετωνικής Προεδρίας έγιναν αρκετές διοικητικές διευθετήσεις ε, ε, σχετικά με την ολοκλήρωση κάποιων αποστολών ε, κοινών με ε, άλλους οργανισμούς όπως ε, ας πούμε με τα Ηνωμένα Έθνη. Οι προσπάθειες ασφάλειας είναι σταθερές όσον αφορά τα όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ε, ε, συζητήθηκαν οι δυνατότητες διασταυρούμενης ε, συνεργασίας με την Αθήνα, το πρόγραμμα Αθήνα. Ένα άλλο ζήτημα δραστηριότητα ήταν η συμφωνία συνεργασίας ανάμεσα στο EDA και τον Μηχανισμό Αθήνα η Λετωνική Προεδρία ε, κινήθηκε έτσι ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας και την ε, Αθήνα που θα, θα μπορούσε να καταλήξει σε ε, πλήρη συνεργασία μεταξύ των δύο και επομένως πλήρη δυνατότητα χρήσης των δυνατοτήτων και των δύο του οργανισμού και του μηχανισμού. Ένα άλλο ζήτημα είναι οι επιπλέον πόροι ε, για τις αποστολές άμυνας και ασφάλειας. Ένα παράδειγμα ε, επιτυχών διαπραγματεύσεων ήταν η μεταφορά ε, κόστους στην, από την κεντρική, στην κεντρική Αφρική προς, του, προς τα Ηνωμένα Έθνη. Τέλος, ε, εγκρίθηκε μια απόφαση σε επίπεδο υπουργικό όσον αφορά τον μηχανισμό Αθήνα ε, έτσι ώστε να ε, υπάρξει καταμερισμός των δαπανών όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό. Πέρα από αυτό πέρα από αυτά τα οποία ε, ανέφερα τώρα, ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε οργανώσει διάφορες ε, στρογγυλές τράπεζες για συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε οργανώσει επίσης ε, κάποια workshops κτλ. Για να ολοκληρώσω τις αρχικές μου παρατηρήσεις, επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που σας παρουσιάζω είναι μονάχα ένα τμήμα των δραστηριοτήτων της Λετωνικής Προεδρίας κατά τη διάρκεια των έξι μηνών ε, έχουμε ως Λετωνική Προεδρία συνδράμει στην καλή λειτουργία όλων των ομάδων που αφορούν θέματα άμυνας και ασφάλειας και θέλω θα με δω ευκαιρίες για να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή. Ε, κινηθήκαμε όλοι και εγώ προσωπικά αλλά και η, υπηρεσία μου ε, υπέρ των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Τώρα, τα μέλη της Επιτροπής μας. Ερωτήσεις. Ο κύριος Κελανο. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ΕΛΚ και της Εστονίας. Είπατε ότι η Λετωνία έχει πετύχει κάποια πρόοδο. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε ε, να εκφράσουμε ικανοποίηση για τη Λετωνική Προεδρία. Το είπατε και εσείς ποια είναι τα επιτεύγματά σας. Είναι σημαντικό να υπάρξει συζήτηση για να ελέγξει τις μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο. Επίσης, χαίρομαι που εμβαθύνεται περισσότερο στη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως θα ήθελα να σας προτείνω να κοιτάξετε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο που είχε εκπονήσει συνάδελφος στην προηγούμενη θητεία, ήδη το 2009. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα βρείτε εκεί μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία και καλές ιδέες. Συνεργασία για την προστασία του κυβερνοχώρου τώρα. Είναι πολύ σημαντικό να οργανωθεί μια τέτοια συνεργασία. Τέλος, για τους υβριδικούς πολέμους. Και αυτό είναι κάτι που χαίρομαι που είναι στην ατζέντα. Τώρα ερώτησή μου είναι, σε αυτό το στάδιο, πώς αξιολογείτε εσείς τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή έχει μπορέσει να πετύχει να έχει μια πιο ενιαία προσέγγιση απέναντι σε αυτούς τους υβριδικούς πολέμους και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ο κύριος Τέτινα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη, επιτρέψτε μου να σας εκφράσω την εκτίμησή μου να σας πω δηλαδή... Να σας πω δηλαδή ότι εκτιμώ πολύ το ρόλο που παίζει η Λετωνία, το ρόλο που έχει παίξει τους τελευταίους μήνες. Έχω μια ερώτηση, ίσως κάπως απλοϊκή. Αναφερθήκατε στη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και την ευάθυνση της συνεργασίας αυτής. Η Λετωνία συμμετέχει στο ΝΑΤΟ Υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο 5 αν δεν απατώμε, τη συνθήκη, που λέει ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να προστατεύει τις χώρες μέλη εφόσον μία χώρα μέλος δεχτεί επίθεση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Το άρθρο αυτό 5 καλύπτει και Μπορείτε να μας πείτε αν το Green Greenman σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε, κύριε Στέτινα. Κύριε Πρέσβη, έχετε συμμετάσχει σε πολλές δραστηριότητες της Λετωνικής Προεδρίας, σε πολλές εκδηλώσεις και θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι υπήρξε, φτιάχτηκε και μια ομάδα φίλων της Προεδρίας. Πολλοί από εμά θα έπρεπε να συμμετάσχουμε. Πάντως η αφοσίεση της λετονικής διπλωματίας των εκπροσώπων ε, όλων πλευρών από τη χώρα, κυβερνητικών και άλλων. Η συμμετοχή τους ήταν μεγάλη. Είχαμε πληροφορίες κάθε φορά που τις ζητούσαμε, οπότε σας ευχαριστούμε. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η δικιά σας εμπειρία για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας, σε αυτό το πόλεμο προπαγάνδας που γίνεται. Επίσης για το κέντρο αριστείας που είναι στη Ρήγα, υπό το Γιάρης Παμπρίξ. Ξέρω ότι αυτό είναι πίτευμα των ε, συναδέρφων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Πάπρικς και άλλων η γνώση όσον αφορά την στρατηγική επικοινωνία, τον πόλεμο προπαγάνδας, είναι πράγματα τα οποία χρησιμοποιούνται για να επηρεαστούν οι πολίτες και οι κοινωνίες στις χώρες μέλη από τη Ρωσία και όχι μόνο από τη Ρωσία. Ο οργανώσεις όπως είναι εκείνη του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, Όλοι αυτοί χρησιμοποιούν τα ίδια μέσα για να μας επηρεάσουν, να επηρεάσουν την νεολαία μας. Στη δικιά σας την ε, Προεδρία θεσμικά πώς είδατε αυτά τα πράγματα, πώς τα αντιμετωπίσατε, μια που μιλάμε και για τη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρω ότι σε πολλές ευκαιρίες έχει τεθεί το ζήτημα, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε προσέξει αρκετά από πλευρά των θεσμικών οργάνων. Χτες μεταξύ άλλων σε μια εκδήλωση ένας από τη ρωσική αντιπολίτευση έκανε την πρόταση να επεκταθούν οι ευρωπαϊκές κυρώσεις, οι δυτικές κυρώσεις, και σε αυτούς που φαίνεται ότι κάνουν την προπαγάνδα, που δεν είναι μόνο δημοσιογράφοι, αυτούς που είναι κοντά στο Κρεμλίνο. Και κατά τη γνώμη μου, είναι πράγματι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος, αν θέλουμε να αποτρέψουμε τη Ρωσία, το Κρεμλίνο να κάνουν τόσο αποτελεσματική προπαγάνδα. Γιατί για να αντιμετωπίσει κανείς αυτού του είδους τον πόλεμο με θετικά μηνύματα και καταδεικνύοντας ότι πρόκειται για χειραγωγία, αυτός ο τρόπος πρέπει να δούμε μάλλον ποιος από τους δύο τρόπους είναι πιο αποτελεσματικός. Για να περάσουμε την κοινή γνώμη. Πάντως πολλά από αυτά τα εργαλεία, όπως είπα, χρησιμοποιούνται και από μη κυβερνητικούς παράγοντες. Είπαμε, είναι από το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος ή από άλλους ριζοσπάστες, ομάδες ριζοσπαστικές που χρησιμοποιούν τρομοκρατικές μεθόδους. Ένα άλλο ερώτημα είναι το εξής. Σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε συζητήσαμε με την Επίτροπο Μπιενκόφσκα. Και ήταν σαφές ότι προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε την αμυντική αγορά στην εσωτερική αγορά. Γιατί όντως υπάρχει θέμα διπλής χρήσης. Ο αμυντικός τομέας Και τα θέματα, έστω και της διπλής χρήσης, δεν είναι θέματα TTIP, όταν μιλάμε για την ασφάλεια και την άμυνα. Έτσι καλώς θα τα συζητήσουμε και αργότερα με εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχουν στο τραπέζι πώς σκεφτόμαστε να λύσουμε το θέμα αυτό της συνεργασίας και στον τομέα αυτό με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ. Κύριε Σαφχάουζερ. Συγγνώμη, πήρα το λόγο κάπως αργά. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Κύριε Πρέσβη, δεν συμμερίζομαι την ανάλυσή σας. Αλλά είναι φυσιολογικό. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω, γιατί και εμένα με ρωτάνε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κοινοβούλιο μας, οι χώρες μέλη, δεν εμπλέκονται περισσότερο στη διαδικασία του Μίνσκ. Δεν βλέπω γιατί αναλύουμε την προπαγάνδα. Κάποιοι θα έλεγα ότι εκφράζουν και ικανοποίηση αν απετύχει αυτή η μοναδική πολιτική λύση. Εγώ ο ίδιος πήγα στο Τόμπασκ 9 Μαΐου. Ήταν σαφές ότι ήταν οι δυνάμεις του Κιέβου που βομβαρδίζανε. Και έρχομαι στις Βρυξέλλες και ξαφνικά μιλούσαν για προδοσία. Όλα δηλαδή στρεβλώνονταν. Λένε οι αρχές ότι πρέπει να αρχίσει η αυτονομία, η αποκέντρωση, που είναι πολύ θετικό. Και το Κίεβο να ελέγχει πλήρως τα σύνορά του οι προτάσεις αυτές έγιναν για μήνες προκειμένου να επιτευχθεί η αποκέντρωση αυτή και δεν ελήφθησαν υπόψη. Μόνο πρόσφατα, επειδή και το Κίεβο εμπλέχτηκε. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το Κίεβο ακούει τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ακούει την Ευρώπη. Οπότε, εσείς γιατί δεν τηρήσατε τις συμφωνίες του Μίνσκ και δεν φροντίσατε για την εφαρμογή τους και γιατί αφήνετε πάντα τους Αμερικανούς να βάζουν μπρος και πάλι τη διαδικασία αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Σαφχάουζερ. Ειλικρινά ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου κάνατε αλλά πρόκειται για ανταλλαγή απόψεων που έχουμε εδώ με τον ε, πρέσβη Πέλς. Με τη Λετωνική Προεδρία δηλαδή. Και δεν θα ήταν, ε, βλέπετε, ευγενικό να μπούμε σε έναν ε, διάλογο εδώ μεταξύ μας. Οπότε, επιτρέψτε μου να ζητήσω από τον πρέσβη να απαντήσει. Εκτός μικροφώνου διάλογος δεν ακούσαμε. Ο πρέσβης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και για όλα τα καλά λόγια που είπατε για την Λετωνική Προεδρία. Πραγματικά χαίρομαι και είμαι υπερήφανος. Θα προσπαθήσω να απαντήσω μία-μία τις ερωτήσεις. Για την ερώτηση του κύριου Κέλαμ, σχετικά με το υβριδικά, με ποιος είναι δηλαδή η προσέγγιση, τι έχει επιτευχθεί και τι θα γίνει στο μέλλον. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει επιτευχθεί την τελευταία περίοδο είναι ότι έχουμε στην ουσία ευαισθητοποίηση για αυτό το υβριδικό ζήτημα που δεν ήταν κάτι που γενικώ ε, ήταν γνωστό ε, σε παγκόσμιο επίπεδο πριν από ένα χρόνο. Οι υβριδικές απειλές είναι ένα αναγνωρισμένο φαινόμενο. Επίσης, από την πλευρά της Προεδρίας, προσπαθήσαμε να βάλουμε στην ημερήσια διάταξη και σε επίσημες και σε ανεπίσημες ε, συναντήσεις, για παράδειγμα μέσα ε, στα πλαίσια της ε, μόνιμης ε, διαρθρωτικής συνεργασίας, το PSC, και μέσα από το έφεση που επίσης γνωμονούμε την είπατε εκπρόσωπο που το έβαλε στη μερίσια διάταξη του Μαΐου και αναφέρθηκαν οι πριδικές απειλές Οπότε έχει αναγνωριστεί το ζήτημα. Το βασικό όμως είναι καταρχάς να δούμε και να κατανοήσουμε τι αυτό σημαίνει για τις εθνικές ε, διοικήσεις σε κάθε περίπτωση. Η Εστονή ήταν πολύ καλή στην αντιμετώπιση αυτού. Είχαμε συναντήσεις με εκπροσώπους από το Τάλιν για αυτό το θέμα. Άρα, κομμάτι της απάντησης στις ηχαφρυδικές απειλές είναι εθνικό. Βέβαια, ε, πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφόρων οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί όπως είπα η διασύνδεση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας γίνεται όλο και πιο θολή. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Αν δείτε λίγο την UNFOR ε, ε, ε, αποστολή που έχει δημιουργηθεί, ένα από τα άτομα που είχε εμπλακεί στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μουσείο του Κάιρο αναφέρθηκε ότι βρέθηκε στην Ιταλία μέσα σε μία από τις βάρκες με πρόσφυγες. Υπάρχει λοιπόν διασύνδεση. Και πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά. Ναι. Μαθαίνουμε λοιπόν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα στις υβριδικές απειλές και μαζί με την Επιτροπή και τις υπηρεσίες της, το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να συνεχίσει να προσπαθεί η δραστηριότητά μας να, να γίνεται σε αυτούς τους τομείς κατά κύριο λόγο και υπάρχουν ε, πολλές ε, δυνατότητες να δούμε πώς θα προχωρήσουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι θα κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Όμως ακόμα ε, τώρα φτάνουμε σε αυτό το σημείο Συμβούλιο. Για αυτό που είπε ο κύριος Στέτινα σχετικά με το άρθρο 5, κατά πόσον λοιπόν αυτές οι υβριδικές απειλές καλύπτονται από το άρθρο 5 ή όχι, η εύκολη απάντηση σε αυτό είναι ότι το ΝΑΤΟ αντιδρά στις απειλές με τον τρόπο του άρθρου 5. Δηλαδή η Βορειοατλαντική Συμμαχία έχει αποφασίσει με αυτόν τον τρόπο να απαντά. Αν το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο, το, το Σώμα των Πρεσβευτών, δηλαδή του ΝΑΤΟ, αποφασίσει ότι θα δράσει έτσι, κατόπιν τίματος κράτους μέλους. Τέλος πάντων, είναι καλή ερώτηση. Δεν θα με ανησυχούσε ιδιαίτερα αν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί γι' αυτό. Εντάξει, ε, μπορείτε να με διορθώσετε, αλλά αυτή είναι η απάντησή μου τώρα. για την ε, ερώτηση της Πρόεδρου, της κυρίας Φατίγκα, για την προπαγάνδα και όλα αυτά. Ναι, είναι πρόβλημα. Καταρχάς να αναγνωρίσουμε ότι η προπαγάνδα δεν είναι δημοσιογραφία. Οπότε πρέπει να δούμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό που είναι δική μας αξία ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην ουσία η ελευθεροτυπία, οι διπλωματικές μας αξίες. Δεν μπορούμε να απλώς να καταργούμε ότι δεν μας αρέσει. Δεν είναι εύκολο αλλά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να, μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. Καταρχάς, έχει αναγνωριστεί ο ζήτημα στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη συμπεράσματα μάλλον, το Φλεβάρι. Αναγνωρίστηκε και στα συμπεράσματα του FSC τον, ε, αργότερα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Μάρτιο έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εντός του Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης μαζί με τα κράτη-μέλη για να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα θα βγει το σχέδιο δράσης Τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, και αυτό είναι και κάποια μαθήματα από το κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ, όπου είναι πρόεδρος ο πρόεδρος Πάτροτ. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι όλα αυτά μπορούμε να τα δείξουμε, να τα αποκαλύψουμε. Δεύτερον, μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες και είναι αλήθεια και κάποιες φορές κατανοητό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας από τους μεγάλους ηγέτες ε, παραφράζοντας τον Νονό είπε ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που όταν σου προσφέρουν κάτι ε, δεν μπορείς να, την να το αρνηθείς αλλά όταν σου κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια προσφορά δεν την καταλαβαίνεις. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει αντίσταση στα μέσα. Δηλαδή ε, υπάρχουν επιρροές από τα κράτη μέσω κονδυλίων. Πρέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επίσης στις κοινωνίες ε, να είναι να υπάρχει στις κοινωνίες επιμόρφωση για το τι είναι ψέμα και τι όχι από όσα αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης πρέπει να δούμε πώς ε, θα εξετάσουμε το θέμα της αγοράς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ε, αυτό είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Την ίδια στιγμή υπάρχουν ξεκάθαρες ε, περιπτώσεις κατάχρησης ε, της εξουσίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης που εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Τώρα για τα ε, προϊόντα διπλής χρήσης και τη συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείε, από όσο γνωρίζω, τα, τα βήματα που γίνονται, ε, γίνονται συγχρονισμένα με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Αν κάνουμε κάτι, ενημερώνονται. Τώρα για το ε, προϊόντα διπλής χρήσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά από περιοριστικά μέτρα αν η συμφωνία του Μίνσκ αποτύχει, και το πει αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο Γενικά, τότε μπορεί να εξετάσουμε την επέκταση των περιοριστικών μέτρων και θα πρέπει. Όμως, σε αυτό το σημείο Και όπως είπε και ο κύριος Σαφχάουζερ, η συμφωνία του Μίνσκ είναι στην ουσία το μόνο πολιτικό εργαλείο που παίζει αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι και πρέπει να το υποστηρίξουμε. Τέλη του έτους είναι ε, η προθεσμία για την εκπλήρωση αυτής της συμφωνίας του Μίνσκ και ελπίζουμε ότι όλα τα μέρη θα συνεργαστούν και θα δουλέψουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, φυσικά θα πρέπει να δούμε αν υπάρξουν και άλλα περιοριστικά μέτρα. Ευχαριστώ. Yes, Mr. once more, please. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρέσβη. Είστε από τη Λετωνία. Ίσως έχετε ακούσει και αυτό που έχει πει και ο Winston Churchill. Όταν υπέγραψε ε, η Ρωσία την ε, ε, συμφωνία ότι από τη στιγμή που υπάρχει υπογραφή έχει αξία το χαρτί. Ε, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό πλέον, ε, γιατί κατά τη γνώμη μου ε, ως τώρα έχουμε δει ότι έχει πεθάνει αυτή η συμφωνία. Προσπαθούμε να δώσουμε επιχειρήματα ώστε να κρατήσουμε τη Ρωσία στη συμφωνία. Μάλλον είναι χαμένη η μάχη, ίσως πρέπει να βρούμε άλλους μεθόδους. Ίσως πιο σκληρές κυρώσεις. Και αυτό ε, θα δείξει στην ουσία ότι είμαστε έτοιμοι να ε, υπερασπιστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες και τη δημοκρατία. Τι περιμένουμε, δεν ξέρω. Thank you very much indeed, uh, Ambassador. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ιδιαίτερα που μας αναλύσατε τα σχέδια προκειμένου να έχουμε νέες επιχειρήσεις. Πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπιστεί και το θέμα των ε, μεταναστών που μας φτάνουν από τη Βόρεια Αφρική ή μέσω της Βόρειας Αφρικής. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι σημαντικές. Αυτό το οποίο μας απασχολεί είναι η ικανότητα πώς ε, μπορούμε να συνεργαστούμε και με άλλους και πώς θα υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για τις προσπάθειές μας αυτές. Προσπάθειες είτε που έχουν ήδη αρχίσει ή που θα αρχίσουν. πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Η σημερινή ε, συνάντηση με τον πρέσβη αφιερώθηκε ακριβώς σε αυτά τα θέματα κυρίως. Όταν μιλάμε για κυρώσεις, είναι γιατί ακούγονται πολλές φωνές τελευταία για τη δυνατότητα να χαλαρώνουν και οι κυρώσεις. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε και πάλι την κατάσταση προς τα τέλη της χρονιάς. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον πρέσβη που ήταν εδώ. Είναι ο πρέσβης μας στην μόνιμη αντιπροσωπεία. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για τη συμμετοχή σας εδώ. Μη φύγετε, θα συνεχίσουμε σε λίγο για το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η συνάντησή μας με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ. Είναι από την αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Λίγα λεπτά διακόπτουμε μόνο.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 Ladies and gentlemen, please be seated. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Συνεχίζουμε με την απογευματική, απογευματινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Ο τίτλος αυτό το σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης είναι η ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στην ασφάλεια και την άμυνα. Θα δούμε την άποψη της Αμερικής. Σύντομα, λοιπόν, μαζί με την αντιπροσωπεία για την συνεργασία ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, αντιπροσωπεία από την αντίστοιχη επιτροπή δηλαδή, έχουμε τον κύριο David McAllister από την ε, επιτροπή, τον οποίο σύντομα θα σας ε, αφήσω να ακούσετε ε, όταν θα κάνει τα εισαγωγικά του σχόλια. Αλλά έχουμε και τους αξιότιμους ε, προσκεκλημένους μας εδώ. Ο κύριος Τζον Σάμις. Ο αναπληρωτής επικεφαλή της αποστολής των ε, Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερο ο κύριος Ρόμπερτ Μπέλ, ο οποίος είναι ο υπεπτός εκπρόσωπος του ε, Υπουργείου Άμυνα και σύμβουλος ε, στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΝΑΤΟ. Καλώς ήρθατε. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο David McAllister. Ευχαριστώ πολύ και ένα θερμό καλωσόρισμα εκ μέρους μου σε όλους σας, αλλά ιδιαίτερα στους αξιότιμους προσκεκλημένους μας. Είναι πραγματικά τιμή μου και χαρά να συμπροεδρεύω αυτή τη συνάντηση για την ενισχυμένη διαδηλαντική συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Η άμυνα και η ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη στην ε, ε, συνάντησε τη δια... Ε, ανα... διακοινοβουλευτική και έχουμε και την επικεφαλής της Επιτροπής ΑΦΕΤ, την πρόεδρο που έχουμε προσκαλέσει. Ας δούμε λίγο πώς γίνεται τα πράγματα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην ευρωπαϊκή γειτονιά μας. Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε γιατί αυτό το θέμα έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στις διατλαντικές συζητήσεις. Γι' αυτό λοιπόν πραγματικά δημονώ να ακούσω πώς οι προσκεκλημένοι μας ε, βλέπουν ε, το ε, πλαίσιο συνεργασίας μέσα στο ΝΑΤΟ αλλά και μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών συγκεκριμένα. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών σε επίπεδο συνεργασίας και εξελίξεων. Αν λοιπόν δεν έχετε ε, πρόβλημα κύριε Σάμιν, να ξεκινήσετε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, ε, David που μας ε, ε, φιλοξενείτε σήμερα εδώ. Η συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ασφάλειας και άμυνας έχει επεκταθεί μέσα στην πάροδο των ετών, όμως ε, χαίρομαι που υπάρχει αυτός ο διάλογος για τη διατλαντική νομοθεσία και περιλαμβάνει την ασφάλεια και την άμυνα στην ημερήσια διάταξη. Η στιγμή η χρονική δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη. Υπάρχουν τεράστιες παγκόσμιες προκλήσεις και χρειάζονται ισχυροί μηχανισμοί συνεργασίας για να τα αντιμετωπίσουμε. Η ομόλογή σας στο Κογκρέσο με χαρά τους έσβησε το μικρόφωνο το μιλητή δυστυχώς. Ε, θα χαρούν να δουν ε, νέε ιδέες για την ενίσχυση της συνεργασίας ε, η οποία θα πρέπει να γίνει πιο ε, αποτελεσματική. Θα σας πω τις απόψεις των ΗΠΑ για μια σειρά από βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, όπου οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη συνεργάζονται. Στις στους πρώτους εννέα μήνες ε, αυτής της κοινοβουλευτικής ε, θητείας είχαμε πολύ σημαντικές επαιτίους. 100 χρόνια από την έναρξη του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 70 από το τέλος ε, του Δεύτερου Παγκοσμίου και 25 από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές ε, θυσίες που έχουν κάνει οι άνθρωποι στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να έχουμε το νέο όραμα της ελευθερίας και της ειρήνης. Η ΕΠΑ είναι αφοσιωμένη σε αυτό το όραμα. Ακόμα και τώρα που υπάρχουν απειλές στην ειρήνη στην Ευρώπη, μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και μια ισχυρή διατηλατική σχέση χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές. Τους πρώτους μήνες που είχαμε τις επιθετικές τάσει της Ρωσίας στην Ουκρανία, ε, βλέπουμε ότι η ελευθερία και η ασφάλεια στην Ευρώπη ανεβαίνει και κατεβαίνει σε σχέση με την Ουκρανία. Πρέπει λοιπόν ε, να δούμε ότι τα τελευταία χρόνια είχαμε μια στεναρή στάση ως προς τις κυρώσεις έναντι ε, της Ρωσίας, όπου την προσπαθούσε να διχάσει τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά δεν το κατάφερε. Ε, θεωρούσε ενδεχομένως ότι εμείς θα ήμασταν υπέρ μιας Ουκρανίας ε, που, διαφορετικής από αυτή που αυτός πρεσβεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 28 ε, μέλη αλλά και οι Ηνωμένε Πολιτείε κατάφεραν ταυτόχρονα σχεδόν να επιβάλλουν τις ίδιες κυρώσεις και αυτό ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα. Πρέπει να κρατήσουμε ψηλά την πίεση ε, δεν πρέπει να σταματήσουμε τις κυρώσεις, πρέπει να τις επεκτείνουμε να συνεχιστεί η επιθετική τάση της Ρωσίας, γιατί είναι εκεί για να υποστηρίξουν τη διπλωματική διαδικασία. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει και να ε, ασκείται πίεση για να εφαρμόσει την συμφωνία του Μίνσκ. Οι κυρώσεις πρέπει να διατηρηθούν μέχρι, πλήρη, μέχρι την πλήρη εφαρμογή της συμφωνία του Μίνσκ, όπω αποφασίστηκε τον Μάρτιο στο Συμβούλιο. Την ίδια στιγμή είναι ανοιχτέ οι πόρτε ε, συνεργασία με τη Ρωσία σε τομείς ε, κοινού συμφέροντος. Θα πρέπει να έχουμε ειρηνική συνεργασία που θα σέβεται την εδαφική κυριαρχία των γειτονικών χωρών. Η Ρωσία πρέπει να είναι ένας υπεύθυνος εταίρος στο διεθνές σύστημα. Μία άλλη βασική προτεραιότητα των ΗΠΑ είναι η συλλογική δράση, ειδικότερα με το, συνεργασία με τους Ευρωπαίους, για να αντιμετωπίσουμε την συνεχή απειλή της τρομοκρατίας, ειδικά από την ε, Αλκάιντα, τον ISIS και τους φίλους τους. Ένας αποφασιστικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτές τις άμεσες απειλές είναι να βοηθήσουμε τους άλλους να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις των σειράξεων και ε, χρειαζόμαστε να ε, έχουμε κοινή προσπάθεια ως προς την αντιμετώπιση της διάθεσης των πυρηνικών ε, όπλων. Επίσης, εργαζόμαστε ως προς την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως η αλλαγή του κλίματος και η λιμώδης νόση. Πρέπει να διασφαλίσουμε όλες τις πτυχές, τον κυβερνοχώρο, το διάστημα, όλους τους επικίνδυνους τομείς και τις απειλές. Επίσης, σε αυτές τις ε, ε, προσπάθειες η συμμαχία μας έχει κεντρικό ρόλο να παίξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες απειλές και να προωθήσουμε την ευημερία στον κόσμο μας που έχει παγκοσμιοποιηθεί. Το 2015 η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας ε, ε, ήταν ένας τρόπος για να επαναδιατυπώσουν οι ΙΠΑ την ε, επιθυμία τους να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικά να γνωρίζουμε τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι προωθεί την ειρήνη και την ευημερία σε όλη την περιφέρεια. Υπάρχουν εκατομμύρια ε, θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσα από την προσπάθεια να γίνει ε, η συμφωνία TTIP και ένα ε, εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού. Επίσης, θέλουμε να εντατικοποιήσουμε την συνεργασία μας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα για πράγματα που ήδη ε, την χάνουν στενή συνεργασία. Ένας τομέας στενού συνοντισμού είναι η ανάπτυξη της ασφάλειας και η πρόληψη των σειράξεων. Το κόστος των σειράξεων στην ουσία μας κάνει ε, να δούμε πόσο κοστίζουν οι ανθρωπιστικές κρίσεις. Ε, θέλουμε να βελτιώσουμε λοιπόν την δυνατότητά μας να προλαμβάνουμε τέτοιες σειράξεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικό της ρόλο να παίξει. Οι μακροπρόθεσμες εξελίξεις και επενδύσεις στην ουσία είναι σημαντικές. Είναι ένας τομέας στον οποίο συντονιζόμαστε στενά και η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη συνεργαστεί στην πρώιμη ειδοποίηση, στην ε, έγκαιρη ειδοποίηση και στην πρόληψη των κρίσεων, ε, έτσι ώστε να υπάρχει σταθεροποίηση και ειρήνευση και όλες οι χώρες να μπουν στο σωστό δρόμο προς τη σωστή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Την περασμένη εβδομάδα Είχαμε τον πρώτο ε, διάλογο που κατέληξε σε επίπεδα ασφάλειας και άμυνας και έχουμε ολοκληρωμένα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε βίες εξτρεμιστικές προσεγγίσεις ε, και να εναρμονίσουμε τις προσπάθειές μας ε, για τις βιοπραγίες και τις σειράξεις. Επίσης, το κράτος δικαίου, η πάταξη της διαφθοράς, η καλή διακυβέρνηση, η πάταξη των εξτρεμισμών και των σειράξεων είναι σημαντικά ζητήματα. Κομμάτι του συντονισμού είναι η πρακτική συνεργασία όσον αφορά στην ε, κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Από την πρώτη αποστολή της ΚΕΠΑ στη Βοσνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΠΑ συνεργάζονται στο πεδίο και με το ΝΑΤΟ και με το Ηνωμένα Έθνη και να αντιμετωπίσουν κοινέ προκλήσεις στα Βαλκάνια, στο Αφγανιστάν, σε όλη την Αφρική και παντού στον κόσμο. Σήμερα η, Πάκε και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν τα, ε, τα πλοία του ναυτικού στην Αφρική και σε άλλες χώρες ε, για να συνεργαστούν και να μπορέσει η διεθνής κοινότητα να καλύπτει ύδατα που έχουν το μέγεθος των ΗΠΑ. Έχουν γίνει πάρα πολλές επιτυχημένες προσπάθειες στο τομέα της πειρατείας. Επίσης έχουμε άμεση συνεργασία με τις αποστολές ε, στο Μπαλί της ΕΚΠΑ, επίσης στη Σομαλία και έχουμε πολλές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ασφάλειας. Για να κλείσω να πω ότι φέτος ε, η ο νομοθετικός διάλογος 27-28 Ιουνίου ε, έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευτυχή στιγμή μετά από το Συμβούλιο ε, στις 25 και 26 Ιουνίου για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας που θα είναι σε κεντρικό σημείο της μερίσιας διάταξης. Έχοντας λοιπόν καλωσορίσει όλα όσα αναφέρθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2013, αναμένουμε τις συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, την επόμενη εβδομάδα για να ε, μπορέσουμε να συμβάλλουμε καλύτερα στην ειρήνη και την ασφάλεια και να συνεργαστούμε καλύτερα με βασικούς εταίρους όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα δίνω το λόγο στο συνάδελφο και φίλο μου, ο οποίος ε, είναι σύμβουλος ε, στον πρέσβη για θέματα άμυνας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, την ε, Συμπρόεδρο γιατί μας ε, κάλεσε σε αυτήν την συζήτηση και να σας συγχαρώ επίσης για την επιλογή του αντικειμένου της συζήτησης εξορισμού. Γνωρίζουμε ότι έχουμε μια πολύ υγιή και καλή συνεργασία ε, ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι γεγονός ότι έχουμε και κοινού στόχους. Έχουμε μια μεγάλη ε, πρωτοφανή ευκαιρία την επόμενη εβδομάδα ε, να επιβεβαιώσουμε για μία ακόμα φορά την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ έχουμε τρία, τρεις, συναντήσεις μέχρι, τρεις συναντήσεις μέχρι τότε. Στα μέσα της εβδομάδας ε, έχουμε την συνάντηση των ε, Υπουργών Άμυνας ε, των χωρών του ΝΑΤΟ και το, την πέμπτη το απόγευμα θα έχουμε 22 ε, υπουργού ε, που Άμυνα από ε, το Συμβούλιο και ταυτόχρονα θα έχουμε και το TRD στην Ρήγα. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντική οργανωτική δουλειά οι δύο πρώτες συνεδρίες κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικές και πολύ καλά διασυνδεδεμένες όχι μόνο γιατί έχουμε τους 22 ε, υπουργούς αλλά γιατί ε, θα έχουμε και την υπατή εκπρόσωπο κυρία Μογκερίνη η οποία θα έρθει ε, στις συνεδρίες του ΝΑΤΟ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή που έχουμε την επόμενη εβδομάδα μέσα από αυτές τις τρεις διασκέψεις να μιλήσουμε με δημιουργικό τρόπο για τον τρόπο με τον οποίο οποίων ε, οραματίζονται ε, την καλύτερη συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οι ηγέτες μας. Βεβαίως ήταν ε, και χθες ένα ισχυρό θέμα στη συνάντηση του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ κ. Στόνεμπεργκ με την ηγεσία της χώρας μου όπου διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει στενότερη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Θα ήθελα να αναφέρω την στενότερη συνεργασία όσον αφορά τον κυβερνοχώρο, καθώς ε, επίσης ε, και την προσέγγιση των διαφόρων μορφών υβριδικού πολέμου. Όσον αφορά την κυβερνοχώρο, τον κυβερνοχώρο ε, έχουμε προχωρήσει ήδη και υπάρχει μια τριγωνική ας πούμε θέση. Οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, και Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ ε, διμερώς και οι δύο πλευρές προσπαθούν να συνεργαστούν για θέματα ε, κυβερνοασφάλειας με το ΝΑΤΟ. Όταν μιλάμε τώρα για υβριδικές μορφές πολέμου δεν είναι τόσο καινούριο στοιχείο γιατί στη διάρκεια της ιστορίας. Is applying that strategy under... Ε, η ασυμμετρική μορφή πολέμου ήταν ε, ήδη γνωστή και οτιδήποτε είναι καινούριο ε, μας απασχολεί και το αντιμετωπίζουμε. Τώρα το σημαντικό είναι ότι κατανοήσαμε ότι πρέπει να έχουμε μία στρατιωτική, οικονομική, διακυβερνητική διάσταση στην απάντηση που θα δώσουμε στις μορφές του υβριδικού πολέμου και μονάχα εάν έχουμε ε, μια στενή σχέση θα μπορέσουμε ε, να προχωρήσουμε από πολιτική άποψη και από την άλλη πλευρά ε, το ΝΑΤΟ μπορεί να δώσει την δυνατότητα έγκαιρης αντίδρασης και ε, επομένως ε, να είμαστε σε θέση μέσω της συνεργασίας αυτής σε πραγματικό χρόνο όταν αντιμετωπίζουμε ε, πραγματικά προβλήματα και πραγματικές κρίσεις να μπορούμε να τις ξεπεράσουμε άμεσα. Εγώ έχω εργαστεί και εργάζομαι και για τον ΝΑΤΟ, εργάζομαι και στην αποστολή των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και μπορώ να σας πω και άλλους τομείς τους οποίους ε, προωθούνται οι σχέσεις ε, συνεργασίας ας πούμε στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό όσον αφορά επίσης την ταυτόχρονη κίνηση προγραμμάτων αμυντικών, ε, όσον αφορά επίσης το Γαλιλαίο, όσον αφορά το CBS, όλα αυτά ε, είναι ε, επίσης η καταπολέμηση της πειρατείας, είναι ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους μπορούμε και συνεργαζόμαστε. Η τρανσατλαντική ε, περιοχή έχει ε, ε, μπει σε μια νέα διάσταση λόγω της Ρωσίας και της επιθετικής της πολιτικής στην Κρυμαία και στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, έχουν αποφασίσει να έχουν παρούσα πραγματική επιχειρησιακή δύναμη, η οποία εκ θα είναι εκεί, βάσει του άρθρου 5 της συνθήκης και οποιαδήποτε, οποιοδήποτε εξωτερικός αντίπαλος αποφασίσει να αναλάβει δράση επιθετική ή παράνομη ε, να μπορεί η απάντηση να είναι άμεση. Βεβαίως συμφωνούμε όταν μιλάμε για συλλογική ε, άμυνα το άρθρο 5 μπορεί να ειναι αμεση βεβαιω συμφωνουμε οταν μιλαμε αμφίσιμο αλλά το ΝΑΤΟ κατέχει μια ιδιαίτερη θέση και η ίδια η συνθήκη λειτουργίας της Λισαβόνας αναγνωρίζει ε, την περίπτωση ένοπλης επίθεσης σε χώρες της Ανατολικής ε, ε, Ευρώπης και επομένως εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε βεβαίως σε ένα σημείο μεγάλης έντασης αλλά παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα αυτά τα οποία ε, θα μπορέσουν να ασκήσουν ε, ε, την δράση της αποτροπής που θέλουμε. Υπάρχουν κατά αναλογία με τους πυλώνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρεις πυλώνες στο ΝΑΤΟ που είναι που ξεκινούν με την απλή ε, αποτροπή ε, και φτάνουν στο ύψιστο επίπεδο που είναι η ατομική πυρηνική αποτροπή. Βεβαίως, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, ε, εμείς ε, με μεγάλη ηρεμία και καθαρότητα πνεύματος ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε και τους τρεις πυλώνες, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην αποτροπή. Πριν από δύο εβδομάδες είχα την τιμή να συνοδεύσω το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ σε μια ε, επίσκεψη που έκανε σε τρεις βάσεις στις νότιες Ηνωμένε ε, Πολιτείες. Επισκέφθηκε μία ε, βάση μαχητικών F-15 και τέτοιου είδους ε, ε, αεροσκάφη βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ρουμανία ε, και, το, και, και αυτή η μονάδα ε, αποτελείται από ε, στρατιωτικούς ε, σε αποστρατεία και παρόλα αυτά εξακολουθούν να ακολουθούν μια εκπαίδευση ιδιαίτερα σημαντική και είναι εξειδικευμένοι κυρίως σε ερευνητικές και ανιχνευτικές αποστολές. Μετά ο Γενικός Γραμματικός Γραμματέας επισκέφθηκε ένα καταδιοκτικό ε, ε, σκάφος ε, το οποίο έχει δυνατότητα πυρηνικής αποτροπής και ε, είναι αυτό το ε, κόρνι το οποίο ε, αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει για την ναυτική βάση της Ουέλγα στην Ισπανία. Επίσης, επισκέφθηκε το υποβρύχιο Αλάσκα και το οποίο μαζί με την υπόλοιπη ναυτική ε, δύναμη θα ξεκινήσει περιπολίες ε, έτσι ώστε να υπάρχει μία πλήρης κάλυψη όλου του φάσματος ε, της αποτροπής. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία της σημαντικής και για τους δυο μας αμοιβές εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Θέλετε μήπως κύριε Μακάλιστερ να αρχίσετε εσείς ή όχι. Α. Τότε παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας και σας κύριε Μπέλ και σας κύριε Σάμις. Όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο το καλύτερο. Αυτό πρέπει να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ, είμαστε ενωμένοι. Οι απειλές βρίσκονται στον Νότο, στις αραβικές χώρες, αλλά και ανατολικά. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι τεράστιες. Νέες προκλήσεις, όπως είπατε και εσείς, ευρυδική πόλεμη, για παράδειγμα, και παντός είδους εξαρτήσεις Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι πρώτα απ' όλα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ανατολική Ευρώπη είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες από τις χώρες που ήταν εξαρτημένες παλιά. Κοιτάξτε, θέλω να πω ότι η διαφθορά έχει χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν και πρόκειται για μια εξάρτηση. Πώς δηλαδή υπήρχε συνεργασία με την Ρωσία. Αυτή ακριβώς η συνεργασία είναι που προκάλεσε διαφθορά στα συστήματά μας. Και ακόμα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες πιέζουν και το πολιτικό επίπεδο να πάρουν αποφάσεις που αντιβαίνουν στη λογική της συνεργασίας δεδομένου των κυρώσεων, και της κοινή αντίδρασης που θέλουμε να έχουμε απέναντι στην ρωσική επίθεση. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει μαζί, μαζί με τις Ηνωμένε Πολιτείε να είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Και όποτε εντοπίζουμε αδυναμίες στο σύστημά μας και κενά, εντάξει δεν έχει άμεση σχέση, αλλά χαίρομαι που οι Ηνωμένε Πολιτείε βοήθησαν στην υπόθεση της FIFA όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Σύστημα από μόνο του δεν ήταν σε θέση. Να, ένα καλό παράδειγμα. Βοήθειας από τις ΗΠΑ που έστειλε το μήνυμα ότι τέτοια διαφθορά είναι μία αποδεκτή. Και το δεύτερο επίπεδο είναι η συνεργασία σε προγράμματα. Υπάρχουν πέντε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα των ΗΠΑ, κάτι το οποίο χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι μας για να μας διχάσουν. Γιατί λένε, να, κοιτάξτε, δεν σας παίρνουν σοβαρά, έχει και δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία και Κροατία. Εγώ χαίρομαι για την πρωτοβουλία των δύο γερουσιαστών για την αλλαγή της νομοθεσίας στις ΗΠΑ. Είναι κάτι που θα το αναφέρω και στη συνάντηση που θα έχουμε στη Ρήγα την επόμενη εβδομάδα. Πάντα εμείς ρωτούσαμε τους συναδέρφους στο Κογκρέσο, αλλά προς το παρόν εκεί δεν έχει γίνει καμία κίνηση. Είμαστε σύμμαχοι, μαχόμαστε κατά της τρομοκρατίας και άλλων προκλήσεων μαζί και πρέπει χωρίς διακρίσεις να αντιμετωπιζόμαστε κι εμείς ως Ευρωπαίοι. Ο κύριος Μακάλιστερ μου είπε ότι προτιμάτε ένας-ένας, μάλλον πρώτα τα διάφορα μέλη της αντιπροσωπείας και μετά απαντήσει. Το κύριο Σπάσκου. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια ερώτηση. Ένα σχόλιο μάλλον και μια ερώτηση. Θα με το μήνυμα γιατί είναι σημαντικό να μεταφερθεί. Βλέπετε, έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για διάλογο εκτός μικροφώνου παρέμβαση που δεν την ακούσαμε. Να αρχίσει και πάλι έλεγα ο διάλογος, ίσως και συνεργασία με τη Ρωσία. Καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι επιθυμητό για διάφορους. Από την άλλη μεριά όμως, το μήνυμα πρέπει να είναι κάποια σημάδια καθησυχασμού. Οι τάσεις που άρχισαν μέσω της στρατηγικής και του προγραμμάτων της Ρωσίας, τι δείχνουν, δείχνουν ότι είμαστε σε μία μακρόχρονη διαδικασία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα συνεχίσει αυτός ο τραγικός καθισχασμός. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πού βάζουμε τα όρια για τα πυρηνικά όπλα. Στο ρωσικό δόγμα είναι ότι πρώτα τα πυρηνικά όπλα θα μπουν στο πεδίο και μετά τα υπόλοιπα όπλα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή τώρα. Δεν έχει πετύχει ακόμα αυτό που ήθελε στην Ουκρανία. Αν Λοιπόν, σκεφτώ ότι η Κρεϊμαία τώρα είναι ρωσική επικράτεια. Δεύτερον, ότι επηρεάζουν μέσω της σύγκρουσης ανατολικά και της αποφάσεις στην Ουκρανία. Και τρίτον, ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει κάποιες δηλώσεις για υποψηφιότητα της Ουκρανίας να γίνει μέλος. Οπότε, αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί να έχει επιθετική στάση η Ρωσία και να θέτει σε κίνδυνο την θέση της και όσον αφορά τις κυρώσεις που μπορεί να χειροτερέψουν, αλλά και τη θέση της στη διεθνή σκηνή. Ή κάνω κάπου λάθος. Και αν κάπου κάνω λάθος στην ανάλυση μου, διορθώστε με παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τέτινα. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερος που είχατε σήμερα το χρόνο να έρθετε εδώ. Στην αρχή μιλήσαμε για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί, οι Αμερικανοί στρατιώτες βοήθησαν την Ευρώπη να απελευθερωθεί και συγκεκριμένα τη χώρα μου, για παράδειγμα. Είμαι από την πρώην Τσεχοσλοβακία και πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκεί και αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Τώρα ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Το 1994 υπογράφτηκε η, σύμβαση, η Συμφωνία της ε, Βουδαπέστης, που ήταν απλή. θα έδινε τα πυρηνικά όπλα η Ουκρανία στην Ρωσία και η Ρωσία δεν θα είχε πλέον εδαφικές απαιτήσει από την Ουκρανία. Η Ρωσία δεν τήρησε αυτή τη συμφωνία διότι κατέκτησε την Κρυμαία και άλλα ε, τμήματα της Ουκρανίας. Ένας από τους εγγυητές αυτής της συμφωνίας ήταν η ΙΠΑ. Απλή ερώτηση τώρα λοιπόν, σε τι βαθμό Λοιπόν, πρέπει οι ΙΠΑ να εφαρμόσουν αυτές τις εγγύησεις. Thank you, Mrs. Anna Gomez. Ευχαριστούμε, κυρία Άννα Γκόμες. Εκτός μικροφώνου, κυρία Γκόμες. Καλώς ήρθατε. Για την Ουκρανία δεν έχω καμία αμφιβολία ότι πρέπει να τηρήσουμε αλλά και να διατηρήσουμε αλλά και να ενισχύσουμε ενδεχομένω τις κυρώσεις. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω εμείς οι Ευρωπαίοι και οι ΙΠΑ συνεργάτες στο ΝΑΤΟ πώς δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε την προπαγάνδα του Πούτιν. Πώς δεν καταφέραμε να εμποδίσουμε την κυβέρνηση της Ουκρανίας ε, να ε, κάνει αυτό το ηλίθιο ε, λάθος και να χρησιμοποιήσει την κομμουνιστικό συμβολισμό το οποίο ωφέλησε τον Πούτιν. Λοιπόν, γενικά η βοήθεια ε, προς την Ουκρανία για την πάταξη της διαφοράς που ήταν μία από τις βασικές επαιτήσεις στο Μαϊντάν και επειδή ξέρουμε που είναι τα χρήματα, τα χρήματα είναι στις δικές μας τράπεζες, στο δικό μας χρηματοπιστωτικό σύστημα, ε, γιατί δεν τα καταφέραμε και εκεί. Βέβαια, έχουμε την άλλη σημαία, το Ιράκ και τη Συρία, που κατέρευσαν ε, γιατί είχαν πατήσει αυτές τις κόκκινες γραμμές με τα χημικές ουσίες που ξαφνικά οι κόκκινες γραμμές είχαν όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Και έτσι θα συνεχίσει. Και εκεί η δουλειά που κάνουμε είναι πολύ κακή. Και δεν καταλαβαίνω, υπάρχει μια συμμαχία εκεί, της οποίας ηγείται η ε, Αμερική με τη βοήθεια κάποιων ευρωπαϊκών ε, χωρών και είναι μια ολόκληρη καταστροφή. 30 τύποι εκεί από το ISIS ε, και κάνουν όλη αυτή τη ζημιά. Τι συμβαίνει. Πραγματικά κριτικάρω τους Ευρωπαίους για τον ανύπαρκτο συντονισμό σε στρατιωτικό αλλά και ανθρωπιστικό επίπεδο και φυσικά το ISIS στο Ιράκ και στην Συρία, το Ισλαμικό κράτος δηλαδή, είναι κρίσιμη σημασία. Υπάρχει ο στρατιωτικός αλλά και ο διπλωματικό ρόλος, γιατί ξέρουμε την Σαουδική Αραβία και άλλους παίχτε που παίζουν ένα άσχημο παιχνίδι εκεί. Η Λιβύη. Ας μην μιλήσουμε για τη Λιβύη, γιατί θεωρώ ότι εκεί είπα έχουν ε, άλλη ευθύνη, αλλά υπάρχουν τεράστιες ε, ανησυχίες σε επίπεδο ασφάλειας. Και όταν σκεφτόμαστε σε επίπεδο τακτικής και στρατηγικής μας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ τι σκεφτόμαστε. Συμφωνώ ότι υπάρχουν στρατηγικές προκλήσεις, ότι έχουμε υβριδικό πόλεμο, κυβερνοασφάλεια, τρομοκρατία. Θεωρώ ότι εσείς, είπα δηλαδή, αλλά και εμείς όλοι, θα πρέπει να είμαστε και ε, αντιμέτωποι με κάποιες παράνομες πράξεις των ΗΠΑ, όπως τη χρήση των μη επανδρομένων αεροσκαφών για να σκοτώνουν κόσμο, αλλά ε, πραγματικά θα πρέπει να συνεργαστούμε γιατί αντιμετωπίζουμε αυτές τις πραγματικέ προκλήσεις. Αυτά πρέπει όμω να διορθωθούν. Τέλος, ε, υπάρχουν στρατηγικέ προκλήσει. Η Κίνα. Πώ βλέπετε την Κίνα. Εγώ είμαι από την Πορτογαλία. Έχουμε κάποιες αεροπορικές βάσεις εκεί που ήταν αμερικανικές και αυτή τη στιγμή η Πορτογάλη, παρόλο που έχει μειώσει την παρουσία της η Αμερική, ε, ε, βέβαια δεν έχει αποσυρθεί πλήρως ε, και ελπίζω να μην γίνει, γιατί δεν είναι κάτι που θέλει η Πορτογαλία. Όμως η Κίνα είναι πολύ ενδιαφέρεται για ένα λιμάνι που είναι κοντά σε αυτές τις αεροπορικές ε, βάσεις, αλλά είναι κάτι παραπάνω από το λιμάνι που τους ενδιαφέρει και κάτι παραπάνω από το εμπόριο. Η Κίνα έχει στρατηγική σκέψη ως προς την παρουσία τους στον Ατλαντικό. Αυτά για την συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτός μικροφώνη, Πρόεδρος, δεν την ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ για τις παρουσίες σας, λέει η κυρία Φωτίκα. Χτες, σε μια εκδήλωση, είχαμε ανθρώπους από την αντιπολίτευση της Ρωσίας, τον κύριο Λέσιος και τον Μιχαήλ Κασιάχνοφ, οι οποίοι μας παρουσίασαν έκθεση του Μπορίς με τίτλο Πούτιν τελεία war. Συγχρόνως υπήρχαν και μέλη του Ατλαντικού Συμβουλίου. Τα συμπεράσματα ήταν περίπου τα ίδια. Συγχρόνως το βράδυ είχαμε μία συζήτηση για μύθους και προπαγάνδα και διαφορές ανάμεσα στη δημοσιογραφία και την προπαγάνδα και το πόλεμο προπαγάνδας. Ακούσαμε πολλές προτάσεις από τη ρωσική αντιπολίτευση και ιδέες και αναρωτιέμαι γιατί όπως πολύ σωστά μας είπατε, η εξολόγηση της προπαγάνδας και η βρυδική πόλεμη είναι κάτι που δεν πρέπει να γνώμε. Υπάρχει ένα κέντρο αριστείας για στρατηγικές επικοινωνίες στη Ρήγα. Αυτό λοιπόν που ζήτησε η ρωσική αντιπολίτευση ήταν να χρησιμοποιούμε πια διαφορετικά εργαλεία για να αποτρέπουμε το Κρεμλίνο από το να χρησιμοποιεί έτσι μαζικά την προπαγάνδα του κατά των κοινωνιών μας. Δεν πρόκειται μόνο για χειραγώγηση, δεν πρόκειται μόνο για το ε, να πούνε την αλήθεια για την κατάσταση, πρέπει να σκεφτούμε και κυρώσει κατά αυτών που οργανώνουν την προπαγάνδα, που δεν είναι δημοσιογράφοι. Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται όλο ιδιαίτερος σε αυτό, στην προπαγάνδα δηλαδή. Να βρούμε τρόπους για να τους αποτρέψουμε. Όχι μόνο να απαντάμε με τον καλό τρόπο, είναι μαζικό και θα πρέπει μαζικά να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τέτοια εργαλεία. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο. Κύριε Μακάλιστερ, εσείς ε, τώρα. Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει άλλος ένας ομιλητής, η Μόνικα Μακοβέη, οπότε κύριε, να την ακούσουμε πρώτα ή θέλετε να πάρετε το λόγο. Ωραία. Πρόκειται για έναν μόνο, έτσι. Κύριε Μακοβέη. Λοιπόν, σας ακούμε, κύριε Μακοβέη. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Μάνικα Μακοβέη και είμαι από τη Ρουμανία. Η Ρουμανία και δημιουργεί ασφάλεια, αλλά και υποφελείται από την ασφάλεια στην περιοχή. Και αυτή είναι η δυνατή της θέση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τη σημασία που δίνατε στη χώρα μου ξέρω ότι βοηθάτε για την σταθερότητα στην Ευρώπη και στην περιοχή. Δεύτερον, οι Ρουμάνοι, και εδώ δεν αναφέρομαι στους πολιτικούς στην εξουσία, οι Ρουμάνοι οι πολίτες χαίρονται για την εταιρική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε ειδική σχέση άμυνα, επενδύσεις και έρευνα. Ένα τρίπτυχο. Θέλουμε να συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτό το δρόμο και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί σας. Τώρα όσον αφορά τη ρωσική προπαγάνδα, γιατί είναι κάτι που ακούστηκε, είναι πολύ επικίνδυνη. Την αφήσαμε για χρόνια. Την αγνοήσαμε για χρόνια. Και ίσως να ξέρετε ότι μεταδίδεται στη γλώσσα των χωρών στις οποίες στάνει η προπαγάνδα αυτή. Και δεν έχουμε το BBC και το Free Europe όπως είχαμε την κομμουνιστική εποχή, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίναμε πιο δημοκρατικές χώρες, ε, σκεφτήκαμε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος και πιστεύαμε ότι είχαμε ελεύθερα μέσα ενημέρωση. Τώρα όμως χρειάζεται πάλι κάτι αντίστοιχο, γιατί όπως σας είπα, το Κρεμλίνο μεταδίδει εκπομπές στις χώρες μας και στις γλώσσες μας. Και δεν έχουμε κάτι, ένα ανεξάρτητο μέσο για να αντιμετωπίσουμε αυτή την προπαγάνδα. Τα εθνικά μέσα ενημέρωσης κατά 90% ανήκουν σε ολιγάρχες και πολιτικούς που έχουν διαφορετικά συμφέροντα πολιτικά ή ακόμα και ποινικά. Συμφωνώ και με την Άννα Μαρία Γκόμες σε ένα βαθμό που ρωτάει οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ πού βρίσκονται. Και δεν είναι τόσο ότι θέλω να ρωτήσω, αλλά θέλω να εκφράσω την ευχή και την επιθυμία η συνεργασία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχυθεί. Βλέπουμε αμερικανικά στρατεύματα, σκάφη και σας ευχαριστούμε σε διάφορες σημαντικές περιοχές και στη Ρουμανία και στη Βαλτική και στη Βουλγαρία, την Πολωνία και η Γαλλία κάποιες τέτοιες χειρονομίες κάνει. Θα ήθελα περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Τώρα για το πόλεμο, μια σκέψη θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Το πρόβλημα τότε δεν είναι το πώς θα υποστηρίξουμε τις χώρες αυτές, αλλά πώς θα τις απελευθερώσουμε. Γιατί συμβαίνει σε λίγες ώρες, ξέρετε, η κατοχή. Δεν θα φτάσουμε όμως σε πόλεμο αν τα μηνύματα που στέλνουμε είναι σαφή, αν έχουμε στρατεύματα, σκάφη και στέλνουμε μηνύματα που λένε μην αγγίζετε. Αυτός είναι ο τρόπος για να αποφύγουμε τον πόλεμο. Το γνωρίζουμε όλοι. Για να κρατήσουμε την ειρήνη πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο ανα πάσα στιγμή. Παρακαλώ. Πολλέ και πλούσιες ερωτήσεις σα. Θα μπορούσαμε να μείνουμε εδώ μέχρι το βράδυ και ακόμα παραπέρα, αλλά δεν γίνεται. Θα έλεγα ο Τζον Σάμις να απαντήσει σε κάποιες από τις ερωτήσεις σας για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα της διαφθοράς, για παράδειγμα, τι γίνεται στο Αμερικανικό Προγκρέσο για την αναθεώρηση όσον αφορά τις πρωτοβουλίες των δύο γερουσιαστών. Και θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για τις δυτικές δημοκρατίες και πώς αυτές μπορούν πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν την προπαγάνδα το τσουνάμι προπαγάνδας. Και ίσως ε, να θες να πεις κάτι εσύ για τη Συρία. Θα μιλήσω και για κάποια στρατιωτικά ζητήματα εγώ ε, και μετά θα σου δώσω το λόγο πάλι. Λοιπόν, στον κύριο Πασκού, να ξεκινήσω με τα πυρηνικά. Συμφωνώ ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη στρατηγική Κάθε σύγχασμου από την πρωτοβουλία που ανέλαβα οι ΗΠΑ σε δισεκατομμύρια δολάρια και, 100, ε, και άλλα 800 εκατομμύρια του χρόνου για... δεν πρέπει να υπάρχει λάθος για το τι θέλουμε να πετύχουμε. Όπως και εσείς έτσι και εμείς ανησυχούμε για το ότι ο κύριος Πούτιν πολύ συχνά αναφέρεται στην πυρηνική απειλή επενδύουν στον εξυγχρονισμό των πυρηνικών, αναπτύσσουν ε, πυρηνικά για λόγους στρατηγικής και παραβιάζουν τη σύμβαση για τον έλεγχο των πυρηνικών που χρόνια μας πήρε να τη φτιάξουμε. Δυστυχώς έχουν μια σκοτεινή πλευρά οι Ρώσοι, δεν είναι κάτι καινούριο για σας. το ξέρετε, υπάρχει κλιμάκωση και αποκλιμάκωση που έχει να κάνει με πυρηνική απειλή. Η στρατηγική είναι ότι παίρνετε κομμάτι γης και ελπίζω δεν μιλάμε εδώ πέρα για χώρες ΝΑΤΟ και μετά επιστρέφεται στο απελευθέρωση άμυνα. Με την απειλή των πυρηνικών, όμως, βάσει του δικού τους του δόγματος, στην κρίση θεωρούν ότι υπάρχει αποκλιμάκωση, αλλά αυτή έχει γίνει με τους όρους της Ρωσίας ευνακούς για εκείνη. Η στρατηγική αυτή έχει βέβαια επιπτώσεις. Εγώ δεν έχω συμπεράσματα να σας πω επ' αυτού, απλώς ότι το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά και το παρακολουθούμε. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορείτε να πείτε ότι η Ρωσία πέτυχε τους στόχους της για πάντα στην Ουκρανία. Όλοι θέλουμε τη διαδικασία που έχει συμφωνηθεί, Μίνσκ. Η συμφωνία του Μίνσκ πρέπει να προχωρήσει, να εφαρμοστεί. Έχει στρατιωτικό και μη στρατιωτικό σκέλος, πολιτικό. Το στρατιωτικό συχνά έχει παραβιαστεί όσον αφορά την εκεχήρια. Δεν έχουν αποσύρει βαριά όπλα. Και πολιτικά θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς η Ουκρανική κυβέρνηση θαραλέα πρότεινε διάφορες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να υπάρξει σοβαρός διάλογος με τους Ρώσους για το που πάει η διαδικασία. Αν όμως το πολιτικό αυτό σκέλος δεν χρησιμοποιηθεί σωστά από τους αποσχιστές και άλλους, τότε ο έλεγχος των συνόρων στο τέλος χρονιάς θα έχει επιβληθεί εκ νέου και η Ουκρανία, όπως κάθε κυρίαρχο κράτος, έχει δικαίωμα να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στην επικράτειά της. Αν δεν πετύχει η συμφωνία του Μίνς, οι δυτικές ε, χώρες θα προχωρήσουν προφανώς σε πιο σκληρές κυρώσεις. Κανείς λοιπόν δεν το περνάει στα ψηλά. Τώρα υπήρχε και κάτι άλλο για τη συμφωνία της Βουδαπέστης του 1994. Για μένα είναι αρκετά προσωπικό πρέπει να σας πω γιατί ήμουν ένας από αυτούς που διαπραγματεύτηκαν το μνημόνιο αυτό του 1994 της Βουδαπέστης. Πήγα πολλές φορές στη Γενέβη, Είχα διάφορες συναντήσεις με Ουκρανούς διπλωμάτες οι οποίοι με ρώτησαν «Μπορούμε να σας έχουμε εμπιστοσύνη» και όταν είπαμε ότι αν εσείς παραιτηθείτε από τα πυρηνικά σας εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα παραβιαστεί η ακερότητά σας, τότε είχε το τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο, μεγαλύτερο από τη Σκίναση ή το Ηνωμένο Βασιλείο εκείνη την εποχή, ο πλωστάσιο. Οπότε και εδώ δεν προσπαθώ να γίνω νομικιστής, ήταν μια πολιτική όμως δέσμευση το μνημόνιο αυτό της Βουδαπέστης. Δεν ήταν νομικά δεσμευτικό, δεν το λέω αυτό για να γλιτώσω τις ευθύνες, αλλά το λέω ως μέλος της Γερουσίας που έχουμε δικαιοδοσία για τις συνθήκες και στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουμε μεγάλη διάκριση ανάμεσα σε δεσμεύσεις που είναι νομικά δεσμευτικές και άλλα που είναι πολιτικές δηλώσεις. Το μνημόνιο της Βουδαπέστης δεν πέρασε από την Γερουσία ως δεσμευτικό. Παρ' όλα αυτά είναι σοβαρό. Και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση Κλίντο το πήρε πάρα πολύ στα σοβαρά και όσοι διαπραγματευτήκαμε τη συμφωνία αυτή το όταν είπαμε στους Ουκρανούς ότι αν είχαν πρόβλημα ε, θα ήμασταν εκεί. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε λοιπόν με την κυβέρνηση Ομπάμα ώστε να βοηθήσουμε πολιτικά, οικονομικά για να τους δείξουμε ότι τηρούμε τις υποχρεώσεις μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ο... Η ίδια η... και Εξωτερικών το είπε. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ πέρα και τις δηλώσεις που έγιναν για το πόσο σημαντικό είναι το μνημόνιο της Βουδαπέστης διάφοροι στην κυβέρνηση Ομπάμα το ξέρουν, δεν έχουν ξεχάσει αυτή τη συμφωνία παρόλο που δεν είναι δυσμευτική. Και τέλος θέλω να τελειώσω και με κάτι ακόμα. Νιάννα αναφέρθηκε στη Ρήγα και στη στρατηγική επικοινωνία. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Είναι πολύ καλή πρόταση. Έχει προταθεί και παλιότερα ε, πριν έχουμε την Ουκρανική κρίση. Και είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται για να καθοριστεί το μέλλον μας. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις άλλες ε, ερωτήσεις που ετέθησαν ε, στις ε, ενδιαφέρουσες αυτές παρουσιάσεις. Ξεκινώντας με το θέμα του, της διαφθοράς, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάποιο διάστημα ήταν οι παγκόσμιοι ηγέτες στην πρόθεση της διαφάνειας, του κράτους δικαίου και τα λοιπά. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε φέρει ε, καλύτερη διακυβέρνηση και καλύτερη ένωμη τάξη στις χώρες ε, που θέλαν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την ε, δράση της και σε χώρες που είναι στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά στην Ουκρανία και σε άλλες χώρες με πρόκληση ως προς αυτό το θέμα της διαφθοράς. Αυτό που έχουμε καταφέρει ως τώρα βέβαια δεν αρκεί, απομένουν πολλά να γίνουν. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να έχουμε διάλογο και έχουμε ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάποιους τομείς και επίσης είναι δίκαιο να πούμε ότι και οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν ε, στην ουσία ρυθμίσει τα δικά τους προβλήματα. Έχουμε διάφορους ε, ε, ηγέτες που έχουν διωχθεί για διαφθορά και άλλες τέτοιες Καλα τέτοια δικαίωμα. Όμως γενικά φαίνεται ότι ο πολιτικός κόσμος έχει προβλήματα σε πολλούς τομείς και πέρυσι ειδικά είχαμε ε, πολύ προωθήσει το διάλογο σε σχέση με το παρελθόν. Πρόσφατα ο κύριο Σούλ, ο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών, είχε έρθει εδώ για τον διάλογο ασφάλειας και άμυνας και συνέχισαν αυτές οι συζητήσεις ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας για τη διαφθορά. Το ίδιο όσον αφορά στις προσπάθειες αντιμετώπισης της προπαγάνδας. Η πλευρά που δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια και έχει και πολλά λεφτά να ρίξει και δυστυχώς ε, υπάρχει και κοινό που δέχεται ε, τα μηνύματά της, έχει μια βραχυπρόθεσμη τακτική. Νομίζω όμως ότι αν ξεκινήσουμε να οργανωνόμαστε ε, επί πρωτοβουλειών όπως οι στρατηγικές επικοινωνίες στην Λετωνία πολλά μπορούν να γίνουν. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε αλλά και στη δική μας κοινωνία έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, υπερβολές. Θα πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε τις δικές μας αξίες, τους θεσμούς που άνοιξαν την επικοινωνία, την ελευθερία του λόγου και τις σημαντικές αξίες που δεν θέλουμε να χάσουμε το πρόγραμμα για την κατάργηση των θεωρήσεων είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα. Δεν θέλω να δείξω έλλειψη σεβασμού σε χώρες που θέλουν να ε, είναι σε στενή σύμμαχη των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους οποίες έχουμε και ιστορικές σχέσεις και δεσμούς. Δεν έχει να κάνει με έλλειψη σεβασμού, λοιπόν. Είναι βέβαια και ε, θέμα τήρησης των απαιτήσεων, των προδιαγραφών, ε, κάτι που όλοι πρέπει να κάνουν. Όσες θέλουν χώρες να έχουν αυτή την ε, κατάργηση θα πρέπει να τηρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Η προστασία αυτού του προγράμματος, αυτού καθεαυτού, είναι επίσης σημαντικό στοιχείο. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, όχι τόσο στην κυβέρνηση, αλλά περισσότερο στο Κογκρέσο, που είναι σκεπτικιστικές θα λέγαμε ως προς αυτό το πρόγραμμα κατάρριξης θεωρήσεων. Ελπίζουμε όμως ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε από αυτό και να υπάρχει πρόοδος. τέλο για το θέμα της Συρίας. Οι ΗΠΑ παραμένουν δεσμευμένε σε μια πολιτική λύση για τη Συρία. Μια νέα κυβέρνηση που δεν θα περιλαμβάνει τον Ασάντ. Προφανώς είναι περίπλοκη η κατάσταση, ειδικότερα με την άνοδο των βίαιων εξτρεμιστών, Αλ-Κάιντα Ισλαμικό κράτος και άλλων και οι Ηνωμένε Πολιτείε και ο συνασπισμός τους συνεργάζονται στενά για να βρουν μια λύση. Η ΙΠΑ ήταν ηγέτης στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και έχουμε μεγάλη αφοσίωση στη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις της σύραξης. Έτσι λοιπόν, ε, να πω κάτι που στο οποίο πραγματικά πιστεύουμε είναι ότι χρειάζεται να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική λύση, ένας διακανονισμός που θα φέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα στο λαό της Συρίας ε, που το αξίζει μετά από την τραγωδία που βίωσε τα τελευταία χρόνια. Yeah. If would you like to follow up? No, I'd be happy to. That that uh, uh, I used to speak Chinese pretty well in Κοιτάξτε, εγώ παλιά μίλαγα κινέζικα, αλλά δεν πάση περιπτώσει να σα πω. Πιστεύω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη ε, έχουν ε, δεσμευτεί ε, να καλωσορίσουν ας πούμε την, ε, τις εξελίξεις ε, στην Κίνα αλλά ε, οι δύο πλευρές επίσης μοιράζονται την ευθύνη για σταθερότητα στην περιοχή. Στην νότια θάλασσα της Κίνας, οπωσδήποτε, μάλλον η νότια θάλασσα της Κίνας, μας δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό και επομένως νομίζω ότι θα πρέπει να ε, επιβεβαιώσουμε και οι δύο πλευρές για μία ακόμα φορά το κράτος δικαίου και την υπερίσχυση της λογικής. Όσον αφορά την κατάσταση στο Ισραήλ, ε, δεν μπορώ να σας δώσω ε, τώρα εξειδικευμένη απάντηση, αλλά πάντως είναι γεγονός ότι σε γενικές γραμμές τα συμφέροντα τα οποία η Κίνα ε, μπορεί να διεκδικήσει σε μία άλλη χώρα όσο γίνονται με σωστό τρόπο και μέσα σε κράτος δικαίου ε, δεν μας ε, δημιουργούν πρόβλημα. Ευχαριστώ. It was pretty exhaustive. Νομίζω, λέει η Πρόεδρος, ότι ήταν πάρα πολύ ήταν εξαιρετικά πλήρης η απαντήση που μας δώσατε. Ίσως ε, μία τελευταία ερώτηση για το Κωσυφοπέδιο, τα Δυτικά Βαλκάνια. Τι, ποιες προσδοκίες έχετε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. το περιβάλλον ε, του ΝΑΤΟ και ο τρόπος με τον οποίο το αντιμετωπίζει το κοσυφοπαίδιο σας είναι γνωστά. Έχουμε επίσης, ε, και το γνωρίζετε εσείς αυτό, ε, την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην χώρα. Βεβαίως ευελπιστούμε επίλυση της κατάστασης Έχουμε μια αποστολή εκεί, η οποία είναι ε, πολύ σημαντική, την ε, λαμβάνουμε υπόψη μας με μεγάλη σοβαρότητα, ε, γίνονται οι απαραίτητες ενδιάμεσες επισκοπήσεις, Παρακολουθούνται όλοι οι κανόνες εμπλοκής που διέπουν την δύναμη που είναι εκεί σταθμευμένη. Έχουμε πραγματικά επενδύσει στο θέμα αυτό ε, και ε, εξακολουθούμε να επενδύουμε μέσα από διασκέψεις τέταρτης γενεάς ε, και από εκκλήσεις έτσι ώστε να καλυφθούν οι υποχρεώσεις βάσει της K4 και ταυτόχρονα Πάντως βλέπουμε ότι εξακολουθεί ε, να υπάρχει αυτός ο βαθμός ε, ε, χρήσης των δυνάμεων που είχαμε και πριν μερικά χρόνια. Όσον αφορά, ξέρετε ότι έχουμε περισσότερο στρατιωτική αρρωγή παρά αποστολή στήριξης. Ε, ευελπιστώ ότι ε, σύντομα ε, θα προχωρήσει με πιο ταχύ ρυθμό η διαδικασία διαλόγου μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου. Ευχαριστώ. Well, the next round of the high-level dialogue will take place on the 20 ο επόμενος, η επόμενη φάση του διαλόγου θα γίνει στις, στην 21η Ιουνίου ε, και βεβαίως φιλοδοξία της Σερβίας είναι να ανοίξει το πρώτο κεφάλαιο ε, όσον αφορά την, την, την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και αυτό είναι σημαντικό νομίζω. Πρόεδρος, εξ ονόματος της ε, Επιτροπής ΣΕΝΤΕ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους έγκριτους ε, καλεσμένους μας ε, για την αναλυτική τους παρουσίαση του, τρόπου των μέσων της αντιμετώπισης που, έχει που έχουν οι Ηνωμένε Πολιτείες όσον αφορά τη συνεργασία για θέματα άμυνας και ασφάλεια ε, βεβαίως εμείς θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον ε, κύριο Μακάλιστερ και τα μέλη της ε, αντιπροσωπείας του για την ενεργή συμμετοχή τους στην συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ. Ναι, και με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται και η συνεδρίαση της Επιτροπής ΣΕΔΕ. 14 Ιουλίου θα είναι η επόμενη συνεδρίασή μας.